των Δημοκρατίας και κράτους δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 135 του κανονισμού. Σύμφωνα με την ε, μέση άταξη θα συζητήσουμε για την ε, Μαλαισία. Θα μιλήσουν πρώτα-πρώτα ε, οι συντάκτες της πρώτης ψηφίσματος. Κορά. Ευχαριστώ, Προέδρο. Οι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζονται κυρίω επί οικονομικών κριτηρίων, λαμβάνοντα υπόψη στα πλαίσια συνοκτική πολιτική το σεβασμό των κανόνων κοινωνικών και περιβάλλοντο συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρονται στο προήμιο τη Συμφωνία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν είναι κάτι δεσμευτικό. Η Μαλαισία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσον αφορά τον αυτόχθονο πληθυσμό και τις μειονότητες έχει μείνει πολύ πίσω και υπάρχουν πάρα πολλές παραβιάσεις. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι μεγάλη ανησυχία των μη κυβερνικών οργανώσεων. Βλέπει την, να δημιουργηθούν διάφορα φράγματα στη χώρα ε, που θα είναι επιζήμια και για τους αυτόχθονους πληθυσμούς και για το περιβάλλον και θα, πρέπει να κατασταθούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και θα πλημμυρίσουν πολλές εκτάσεις που τώρα είναι τροπικά δάση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, διαφθοράς. Ε, γίνεται μεγάλη κερδοσκοπία πλευρά των ξενοπενδυτών. Σύμφωνα με ΜΚΟ, 80% των δασών έχουν καταστραφεί για ε, την αφιτευτούν φοινικέ, την παραγωγή φοινικέλαιο. Είναι η Μαλαισία η πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο. χρησιμοποιήσουμε το μέσο των συμφωνίων ελευθέρων συναλλαγών για να ενισχύσουμε αυτή την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι αυτή πιστεύω ότι είναι η ευκαιρία μας. Ευχαριστώ κύριε Κοράο. Συνάδελφε σμάκερ, για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Μαλαισία ολισθαίνει προς ένα αυταρχικό κράτος. Σήμερα είναι επικίνδυνο να διαδηλώνει ειρηνικά και να φοράζει για παράδειγμα ένα κίτρινο μπλουζάκι. Το χρώμα θεωρείται συνώνυμο ισχά της προδοσίας. Τόσος φόβος πια για τη δημοκρατία είναι κακό ιονός. Το εθνικό μέτωπο, η Μπαρισάν Νασιονάλ όπως λέγεται, ε, κυβερνάει εδώ και 58 χρόνια, αλλά ε, βασίζεται σε αρχαϊκούς ε, απικιακούς νόμους. Η ελευθεροτυπία και η ελεύθερη έκφραση πολύ εύκολα περιστέλλονται. Βασίζεται στη σαρία τα νομοσχέδια. Δεν έχει δηλώσει η Μαλαισία ότι θέλει να βοηθήσει και να προβληθεί ως μετριοπαθές Ισλαμική ως μειοτροπαθή Ισλαμική χώρα που καταπολεμά τον Ισλαμισμό. Τι γίνεται με τις μειονότητες. Οι αυτόχθονες όπως η Οράν Ασλή ε, έχουν ακόμα προβλήματα με τα δικαιώματά τους και στην κυριότητα και στην ιδιοκτησία. Ε, καλό το ε, τον Πρωθυπουργό να ε, σέβεται την ε, κοινοβουλευτική δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα λάβει όλα αυτά υπόψη της στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες. Η κυρία Λόχ Μπίλερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μαλαισία οι περιοριστικοί νόμοι χρησιμοποιούνται για να περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης και του διαδηλών μαζικά. Κυρίως η κοινωνία των πολιτών που εκφράζεται επικριτικά κατά της κυβέρνησης κινδυνεύει να συλλαμβάνεται. Και είναι πολιτικές οι προφανώς. Οι κριτικές φωνές ε, ε, βρίσκουν απέναντί τους ε, καταγγελίες και μηνύσεις. Υπάρχει ο νόμος ε, περί ανταρσίας του 1948 Sedition Act που είναι επί απεικιοκρατίας. 40 άτομα ανακρίθηκαν, ε, κατηγορήθηκαν ήδη ε, φέτος ή ε, συνελήφθησαν. Ο Χαλίτης Ματ τον Οκτώβριο δικάστηκε βάσει του νόμου περί επικοινωνίας και περί ανταρσίας διότι δημοσίευε κάποια πράγματα για την κατάχρηση εξουσίας. Ο κόσμος συλλαμβάνεται αυθαίρετα ε, όπως και ο Ράσαν, ο οποίος ε, συνελήφθη το Σεπτέμβριο διότι ε, κατήγγειλε τη διαφθορά ενός κρατικού επενδυτικού οργανισμού. Γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση να αφήσει ελεύθερους και να εγκαταλείψει όλες τις κατηγορίες εκείνων που διαμαρτύρονται ειρηνικά και χρησιμοποιούν το δικαίωμα του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε και θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν και να καταργηθούν τελείως αυτοί οι νόμοι. Το Δεκέμβριο αποφασίστηκε και ένας νόμος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για περιττέρου περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλη συντάκτη των προτάσεων ψηφίσματος. Η κυρία Βίκστρομ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτές είναι οι εξελίξεις στην Μαλαισία. Έχουμε ε, την περιστολή των δικαιωμάτων και βασικών ε, δημοκρατικών ελευθεριών. Οπότε κάνει ό,τι μπορεί για να δημόσει τους επικριτές η κυβέρνηση. Ε, και, και πρέπει εμείς να καταδικάσουμε αυτά τα γεγονότα. Η κατάσταση των δικαιωμάτων στη χώρα αυτή είναι πάρα πολύ κακή και σύμφωνα με την νομοθεσία η κοινωνία των πολιτών, οι πανεπιστημιακοί, τα ΜΜΕ και η αντιπολίτευση υφίστανται επιθέσεις. Γι' αυτό και απευθύνουμε έκκληση μέσω αυτού του ψηφίσματος να αποφυλακιστούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Θα πρέπει ο κόσμος να έχει ελευθερία έκφρασης. Όμως αυτό την σήμερα ημέρα είναι ε, ένας κίνδυνος. Θα πρέπει επομένως να σταματήσουν οι διώξεις και η άσκηση βίας για τους ΛΟΑΔ στη χώρα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθεί το σχετικό ψήφισμα για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι η ελευθερία έκφρασης και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να περιστέλλονται καθιονδήποτε τρόπο. Είναι σημαντικό καθήκον αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και εδώ και παντού. Άλλο συντάκτης του ψηφίσματος λέναρς. Ένα λεπτό στα αγγλικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με το σημερινό ψήφισμα διατρανώνουμε και πάλι ε, ε, τη συμπαράστασή μας στο λαό της Μαλαισίας και τη φιλία μας. Και γι' αυτό ανησυχούμε και έχουμε θορυβηθεί πάρα πολύ για το νόμο περί ανταρσίας που είχε δεσμευτεί να καταργήσει, να ακυρώσει η Μαλαισία. Το αντίθετο έκανε, τον ενίσχυσε. Και ο νόμος για την ασφάλεια εγκρίθηκε χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Δίνει ευρύτατες ε, εξουσίες στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για να επιβάλλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γενικά ανησυχούμε για την ατμόσφαιρα που επικρατεί και αφορά ε, την κοινωνία των πολιτών, τους αντιφρονούδες την αντιπολίτευση και τους δημοσιογράφους. Μεγάλες δυσκολίες έχουν να λειτουργήσουν δεν τα κάνουμε όλα αυτά επειδή μας αρέσει να επικρίνουμε τη Μαλαισία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα και θα πρέπει να λέγονται όλα αυτά. Και από εκεί να αρχίσει ένας επικοδομητικός διάλογος και με τη Μαλαισία και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στις διμερείς μας σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαλαισία, ειδικά τη στιγμή που συσφίγουμε τις σχέσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και η κυρία Βερζά είναι συντάκτρια του κειμένου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Βάριν Μπριμ είναι ένα σύμβολο φιλελεύθερος που έπεσε, προσπάθησε να χειριστεί την κρίση του τέλος δεκαετία του 90. Επέβαλε λιτότητα σκληρότατη, αλλά επίσης ακύρωσε και μεγάλα βιομηχανικά έργα τα οποία δεν ήταν διαφανή. Αφόρητα σε μια χώρα που η διαφθορά κυριαρχεί. Δημιούργησε το Παταϊκάν Χαϊάτ, ε, προσπαθώντας να γεφυρώσει τις διαφορές τις κοινοτικές. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση τελικά ε, οδηγόταν στη φυλακή ε, λοιπόν, και ήταν για θέμα ηθών. Λοιπόν, ε, καταπιέζονται διάφορες μενότητες των ΛΟΑΔ, των γυναικών, είναι τα πρώτα αλλά και δημοσιογράφοι, διανοούμενοι, ε, μαχητές των διαφόρων κινημάτων. Υπάρχει μεγάλη καταπίεση και η εξουσία χρησιμοποιεί μεγάλη βία για να διαφυλάξει τα συμφέροντα της ελίτ. Χρειάζεται καλύτερη ανακατονομή του πλούτου και πολιτικός διάλογος με όλες τις συνιστώσεις. Μόνο έτσι θα βγει η χώρα από τα αδιέξοδο. Χρησιμοποιώντας τα σκεφτικά θέματα με τον κίνδυνο να φτάσει σε ακρεφνείς θέσεις τι σκεφτικές. Άρα πρέπει να δράσουμε γρήγορα για να μην βυθιστεί σε αυτό τον εξτρεμισμό. Ευχαριστώ, συνάδελφε Παντσέρη που έχετε ετοιμάσει την πρόταση ψηφίσματο. για το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στη Μαλαισία είδαμε ότι υπάρχει μεγάλος περιορισμός της ελευθερίας του λόγου λόγω των νόμων που προσπαθούν να κάνουν να σιωπήσουν οι επικριτικέ φωνές. Ανησυχεί ιδιαίτερα ο νόμος όσον αφορά ε, την αντίδραση που, ε, που ε, για αυτό το λόγο το 2015 συνέχισαν πάνω από 100. Ο κ. Ιμπραήμ καταδικάστηκε ε, για Λοιπόν, ε, λοιπόν, και ο σκητσογράφος Ουλάκ επίσης κατηγορήθηκε σύμφωνα με τον νόμο για, ε, μεγάλη, για αντίδραση έναντι της κυβερνήσεως και καταδικάστηκε όπως και η Ιμπραήμ. Τα μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυξανόμενες όσον αφορά ε, την αναφορά, την προβολή των κατηγοριών για διαφθορά εναντίον του Πρωθυπουργού και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τους ΛΟΑΔ. Λοιπόν, ε, και είναι πρόεδρος του ΑΖΕΑΝ η Μαλαισία και είναι σαφές το αίτημα του Κοινοβουλίου να απελευθερωθούν οι καταδικασμένοι να και ε, θα πρέπει λοιπόν να, να ελεγχθούν και οι εξουσίες που έχει ο Πρωθυπουργό. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ διαφυλάξεως της ασφάλειας εθνικής και να προστατεύονται και τα διάφορα πολιτικά δικαιώματα και δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Ας ακούσουμε κάποιες παρεμβάσεις των πολιτικών ομάδων για το Λαϊκό Κόμμα Συνάδελφοι Κέλλη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εργάζομαι στην προσωπία τη σχέση με την Μαλαισία και γιατί επιδεινώνεται η σχέση μα με τη χώρα αυτή. Γιατί ε, είδατε τι έγινε στη συνάντηση τη ε, Σιγκαπούρη για τι εμπορικέ σχέσει. Και βέβαια βελτιώνονται οι εμπορικέ σχέσει, αλλά από την άλλη μεριά οι ευκαιρίε στην χώρα για να υπάρξει ελευθερία έκφρασης και λόγου συνεχώς μειώνονται και μας ανησυχεί ιδιαιτέρω το ότι ε, αυτοί οι νόμοι καταστολή αντί να καταργηθούν συνεχίζουν να ισχύουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για την ελευθερία της έκφρασης. Μια σειρά προσώπων έχουν ε, υποστεί έρευνες, σύλληψη και παραμονή στη δικαιοσύνη. αυτό είναι απαράδεκτο Επίσης ε, βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας η χώρα και η μεταχείριση των ΛΟΑΔ είναι επίσης απαράδεκτη. Μια που όλοι βαδίζουν προς αντίθετη κατεύθυνση και στη δική μου χώρα ακόμα. Ε, είναι απαράδεκτο να καταπατώνται έτσι ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πηγαίνουν σε αντίθετη κατεύθυνση από εμά οι εμπορικοί μα εταιρεία. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη σχέση μα με την Μαλαισία. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη, λέει ο πρόεδρο, για 1,5 λεπτό για του σοσιαλιστέ δημοκράτε. Θα έχει το λόγο η κυρία Γκίλ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και κύριε επίτροπε. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την ε, χώρα πρόσφατα και με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι αυτά τα οποία μαθαίνουμε για την χώρα δεν έχουν μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Είναι σύγχρονη και δυναμική η χώρα. Όμως κάτω από αυτή την επιφάνεια της ε, δυτικόστροφης ε, οικονομίας βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο γίνεται αυταρχική η διακυβέρνηση και δεν μπορεί να μιλήσει κανείς ελεύθερα. Και πάρα πολλοί ε, σύμφωνα με αυτό το νόμο Sedition Act παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα τα οποία δίνουν υπερβολικές εξουσίες στις διοικητικές αρχές, στον ε, Πρωθυπουργό και η καταστολή βασιλεύει. Και ε, όπως ξέρουμε το Σεπτέμβριο έγινε εκείνη η διάσκεψη κατά της ε, διαφθοράς και τότε ρώτησα τον Πρωθυπουργό γιατί εσείς δεν κάνετε κάποιες έρευνες με διαφάνεια για αυτές τις ε, κατηγορίες ε, διαφθοράς εις βάρος σας, γιατί δεν αφήνετε τον κόσμο ειρηνικά να διτυπώσει τις απόψεις του και να κατέβει στο πεζοδρόμιο, γιατί δεν ε, τηρείτε την υπόσχεση να καταργήσετε αυτά τα, αυτούς τους νόμους καταστολής και να μην συνεχίσετε την πολιτική καταστολή, να έχετε διάλογο στην κοινωνία των πολιτών, να απελευθερώσετε τον ε, Ιμπραήμ, τον Ανουάρ Ιμπραήμ και θα πρέπει η χώρα να γίνει ένας ε, φάρος δημοκρατίας. Οι αρχές της ε, χώρας, από ό,τι φαίνεται, φοβούνται ότι αν κάνουν όλα αυτά που τους προτείνουμε θα αποδυναμώσει θέση τους. Όμως το αντίθετο ισχύει. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μαρίνιο Πίντο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Οι σχέσεις, ε, ή μάλλον οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μαλαισία όπω και σε πολλέ χώρε του κόσμου γίνονται μέσα από ένα σύστημα δικαστικό που είναι άκρως διεφθαρμένο. Υπάρχουν νόμοι ε, φρικτοί όπως ο νόμος περί ανταρσίας Sedition Act και ε, χρησιμοποιεί ε, το κράτος, η κυβέρνηση, τα δικαστήρια για να ε, διώκει, να καταδιώκει και να καταδικάζει τους αντιφρονώντες. Πάνω από χίλιοι είναι οι πολίτες που περιμένουν στις φυλακές της Μαλαισίας να τους επιβληθεί η θανατική ποινή. Να εκτελεστεί δηλαδή, γιατί είναι ήδη κατάδικη. Θα πρέπει ε, να τα καταδικάζουμε όλα αυτά και να τα καταγγείλουμε με οικονομικές κυρώσεις όπως το πάγωμα των εμπορικών συμφωνιών που έχουμε με τη χώρα αυτή και ενίσχυση του Διεθνές Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτά είναι όλα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να διατρανώσουμε στη Μαλαισία ότι η παραβίαση των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών δεν ε, μπορούν να παραμείνουν ατιμόρυτα διότι έχουν και συνέπειες οι πράξεις και οι παραλήψεις μας θα πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν να έρθουν ενώπιον του διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Μία εγγεγραμμένη ο κύριος Φουντούλης, παρακαλώ, για 1,5 λεπτό. Η κατάσταση στη Μαλαισία δεν χωράει αμφιβολία πως δεν είναι καθόλου καλή και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες όπως ο καθένας μας τις αντιλαμβάνεται. Πράγματι η Μαλαισία εξελίσσεται πολύ γρήγορα σε ένα αστυνομικό κράτος με περιορισμένη ελευθερία της έκφρασης πολιτικές διώξεις και κατασκευασμένες κατηγορίες. επιπλέον η διαφθορά λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις. σε κάθε περίπτωση όμως κανείς δεν έχει ορίσει την ένωση παγκόσμιο επιτηρητή ούτε της έχει δώσει την εξουσία να παρεμβαίνει και μάλιστα τόσο απροκάλυπτα στα εσωτερικά τρίτων ανεξαρτήτων κρατών. ούτε κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια ούτε μπορούμε να πούμε πως όλα αυτά δεν συμβαίνουν στις χώρες της ευρώπης πολιτικές διώξεις έχουμε κατηγορίες κατασκευασμένες και κατευθυνόμενες κατά πολιτικών αντιπάλων έχουμε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη έχουμε ψευδομάρτυρες σε αυθονία διαθέτουμε και αντίστοιχα ασυλία ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός. όσο για τη διαφθορά κάθε λίγους μήνες έχουμε και ένα καινούριο σκάνδαλο στην ευρώπη με εξαφανισμένα χρήματα αδήλωτα και δωράκια από μεγάλες εταιρείες. οπότε θεωρώ πως πάει πολύ να κουνάμε το δάχτυλο σε ολόκληρο τον κόσμο προσκολλημένοι ακόμα σε κοιοκρατικά συμπλέγματα χωρίς ειδικά να έχουμε πρώτα βάλει τάξη στα του οίκου μας. τέλος αν όντως θέλουμε να πιέσουμε τη μαλαισία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες ας δοκιμάσουμε έναν άλλο τρόπο ας διακόψουμε κάθε εμπορική επαφή με το συγκεκριμένο κράτος κάθε οικονομική ενίσχυση μιας και υπάρχουν διεφθαρμένοι πολιτικοί αξιωματούχοι όπως λέτε και ελοχεύει ο κίνδυνος να οικειοποιηθούν τα χρήματα και ας απαγορεύσουμε στις μεγάλες ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρείες οποιασδήποτε δραστηριότητα σε εκείνη τη χώρα αν έχουμε το σθένος. διαφορετικά κρατήστε την υποκρισία σας εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. σας ευχαριστώ. κύριε Φουντούλη, κύριε Σταραμπέλα, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Μάρκα, έχεις το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ενώ η Μαλαισία είναι μια χώρα με ταχεία και εντυπωσιακή ανάπτυξη και μοντέλο και πρότυπο για την νοτιοανατολική ανατολικη Ασία, πώ μπορεί να παραμένει αγκιστρωμένη σε πρακτικέ του παρελθόντο, βασανιστήρια και θανατική ποινή. Παρόλο που έχει υπογράψει πολλέ διεθνεί συμβάσει, ε, διαπιστώνουμε με λύπη μα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι προτεραιότητα και μάλιστα έχουν πιστοδρομήσει. Θυμίζω ότι συμμετέχει στι 58 χώρε που ακόμα δεν έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Και επίση ε, με 18 χώρες που καταψήφισαν το δικαιοστάσιο μορατόριο για τη θανατική ποινή στις 18 Δεκεμβρίου 2014 στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενική Συνέλευση. Ε, ε, και δεν υπερψήφισαν ε, και ψήφισαν αποχή κάποια άλλη. Γιατί δεν μπορούσε η Μαλαισία να προχωρήσει στις εμελιώδεις ελευθερίες των πολίτων. Ο πρόεδρος. Κύριε Ταραμπέλα, υπάρχει με ερώτηση για σας. Από πλευράς ε, του συναδέλφου Τσερνέσκη, δεχόσαστε. Συνάδελφε Τσερνέσκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Ταραμπελά και τον ευχαριστώ που δέχθηκε ε, την ερώτησή μου. Νομίζω ότι ε, ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο. Αλλά για το συγκεκριμένο θέλω να σας ρωτήσω. Κάτι που ρωτώ συχνά εδώ μέσα. Μήπως θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτές τις προσπάθειες περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ασκηθεί οικονομική πίεση προς τις χώρες αυτές που παραβιάζουν τα βασικά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τι πιστεύετε, απάντησε κύριο Σταραπελά. Συμφωνώ πολύτως με την ανησυχία σας κύριε Τσαρνέσκη, κύριε Αντιπρόεδρε του Κοινοβουλίου επανειλημμένα όταν μιλούμε για θέσεις και ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, το λέμε αυτό, ότι θα πρέπει να γίνει πρόοδος ανθρώπινα δικαιώματα και το κάνουμε προς όλες τις χώρες. Παράδειγμα προς την Κολομβία, που ήταν ιδιάζουσα η κατάσταση. Θυμάστε ότι οι μισοί συνδικαλιστές που ε, δολοφονούνται τον κόσμο είναι από την Κολομβία και στην Κολομβία. Ε, θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι δεν υπάρχει ισότητα εδώ. Πρώτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά η business και όχι το αντίστροφο. Ευχαριστώ και Ταραμπέλα. Ξεκινάει η διαδικασία του Catch the Eye. Συνάδελφε, πώς πισήλ έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ζητούν προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μαλαισία καταβάλω και εγώ προσπάθεια τον τομέα. το κράτος δικαίου δεν ισχύει εκεί, σε αυτή τη χώρα. Και το νομοσχέδιο περιστάσεις χρονολογείται από το 48. Ε, γυμνώνται εύκολα διώξεις ανθρώπων για τα πάντα. Πολύ πρόσφατα το συνταγματικό δικαστήριο απεφάνθη ότι ε, ο νόμος ε, συνάδει με το, με το Σύνταγμα και ο ποινικό κώδικας ε, είναι πολύ αυστηρός. Χίλιοι άνθρωποι περιμένουν εκτέλεση στι φυλακέ. Γι' αυτό, Επίτροπε, υποστηρίζω όλα όσα ανέφεραν συνάδελφοι. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και να συνεννοηθούμε με την ε, Μαλαισία. Αυτό είναι σαφέ, Αλλά οι συμφωνίε μα θα πρέπει να συνάπτονται με τη χώρα αυτή όταν καταργηθούν αυτοί οι νόμοι που δεν κάνουν αυτή τη χώρα να είναι μια χώρα με το κάτω δικαίου. Επόμενο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η έλλειψη ελευθερίας της έκφρασης η θρησκευτική καταπίεση οι διακρίσεις σε βάρος των αυτόχθονων πληθυσμών και των μεταναστών στη μαλαισία είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. η μαλαισιανή κυβέρνηση με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας συλλαμβάνει και φυλακίζει επαόριστον οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται δίθεν ύποπτο για λόγους εθνικής ασφάλειας ενώ οι συλλήψεις εκείνων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι συχνές. επιπλέον η κυβέρνηση της χώρας έχει επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και γι' αυτό έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις χώρες με το χειρότερο βαθμό στην ελευθερία της έκφρασης μια χώρα όπου εφαρμόζεται η σαρία. οι περιπτώσεις όπου οι μαλαισιανές αρχές έχουν επιβάλει κυρώσεις για δημοσιεύματα που εναντιώνονται στην κυβέρνηση είναι πολλές. απέναντι στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη μαλαισία η ευρωπαϊκή ένωση καλείται να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση της χώρας προκειμένου να καταργήσει τον νόμο περί ανταρσίας και να κατοχυρώσει τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης του συνέρχεστε και όσα στηρίζονται στο διεθνές σύμφωνο ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σόγκορ και εσείς ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ε, στη συζήτηση ε, ε, σε κάτι που υπόθηκε χτες ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα και να λογοδοτούν οι χώρες για την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό τους. Και στην ιστορία της Μαλαισίας επανειλημμένα έχουμε δει τέτοια φαινόμενα. Ε, ο κύριος Ιμπραήμ υφίσταται ιδιαίτερη ε, δίωξη. Ε, και ε, μάλιστα τον έχουν κατηγορήσει για σοδομισμό. Ε, το κοινοβούλιο και μάλλον η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει ελεύθερες εκλογές. Είναι η κατάσταση τραγική και η αντιπολίτευση καταστέλλεται. Εμείς προφανώς δεν μπορούμε να ε, αναμειχθούμε στα εσωτερικά της, αλλά μπορούμε να εκφράσουμε τη δυσφορία μας και ε, να επιμείνουμε. Ευχαριστώ, Καστάλτο. Και εσείς ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Καστάλτο. Αυτά, αυτά όλα τα νομοθετήματα. Έχουμε ένα, μια ολόκληρη σειρά από νομοθετήματα αλλά και τον νέο ποινικό κώδικα που χτυπάνε την ελευθερία έκφρασης και ελευθερία του συναθρίζεστη. Ατέλειωσε αυτός ο κατάλογο γίνεται κοινωνικό ντάμπινγκ. υπάρχει μέχρι την ανώτατη πέρα της κυβέρνησης διαφθορά και πρόκειται για επίσης ε, χειραγώγηση από τους πολιτικούς της δικαιοσύνη. Αλλά επίση χειραγούνται και οι δημοσιογράφοι ε, και επίση και ο Αμουάρ ε, Ιμπραήμ ε, φυλακίστηκε για κάποια γελία ε, κατηγορία. Οπότε βλέπουμε πώς εφαρμόζεται η Σαρία και καταστρέφεται το περιβάλλον σύμφωνα με τα όσα είπε προηγουμένως και ο συνάδελφος Κοράου. Είμαστε υπερδύναμοι οικονομική και συνεχίζουμε και έχουμε εμπορικές συμφωνίες αλλά αυτές οι συμφωνίες ε, μπορεί να είναι όπλο για να γίνουμε και υπερδύναμοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα θα πρέπει να μην ε, ενεργούμε ανεξάρτητα από αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους ε, εταίρους μας. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχουμε αυτή τη συζήτηση με αυτό το ψήφισμα. Όλα αυτά αποτελούν κομμάτι των σχέσεων με αυτό, αυτή μας τη χώρα που είναι εταίρος και όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές θέλω και εγώ να επισημάνω πώς έχουν τα πράγματα για την κατάσταση του κράτους δικαίου γιατί θα έπρεπε η συμφωνία με τη χώρα αυτή να έχει ως προϋπόθεση την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα γι' αυτό και νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να πιέσει, θα πρέπει στα σοβαρά να εφαρμόσει την αιρεσιμότητα για τις εμπορικές σχέσεις και με τη Μαλαισία και έτσι να βελτιωθεί η κατάσταση των δικαιωμάτων στη χώρα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σβόμποντα. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Βέντα. Είναι όμως εδώ. Δεν τον βλέπω στη θέση του, αλλά ζήτησε το λόγο. Α, τότε το Καζιδιά τελειώνει σε αυτό το σημείο. Θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Στυλιανίδη και το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Μαλαισία έχει σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Νοτιοανατολική Ασία. Η Μαλαισία έχει την Προεδρία της ΑΖΕΑΝ σε μια εποχή όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για τη δημιουργία μιας οικονομικής κοινότητας ΑΖΕΑΝ. Οι διμερείς μας δεσμοί έχουν ενισχυθεί σημαντικά μέσω αυξήσεως του εμπορίου και των επενδύσεων, μέσω πολιτικού διαλόγου και μέσω πολλαπλών δραστηριοτήτων συνεργασίας. Παρά το γεγονός αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για κάποιες από τις εξελίξεις στη χώρα που έχουν λάβει η χώρα μετά το 2014 εξελίξεις που έχουν πλήξει την ελευθερία της έκφρασης και το κράτος δικαίου. Ανησυχούμε όλος ιδιαίτερος για την αύξηση της χρήσης του νόμου περιστάσεως όπως αποκαλείται και ανησυχούμε η δικαστική απόφαση που αφορά τον κύριο Ανουάρ Ιμπραχήμ που είναι ηγέτης της αντιπολιτεύσης Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, ανησυχούμε επίσης. Θα θυμόσαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη λύπη της για την αυξανόμενη χρήση από το 2014 και μετά της, του νόμου περιστάσεις παρά την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα ανασταλεί αυτός ο νόμος. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να επενθυμίσω ότι τον Απρίλιο του 2015 η ύπατη εκπρόσωπος εξέφρασε δημοσία ανησυχίες ότι αυτό θα είχε συνέπειες για την ελευθερία της έκφρασης. Η ότι εκπρόσωπος εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη σωστή ε, εφαρμογή του νόμου μετά από την καταδίκη του Μοσχοδικού Δικαστήριου της Μαλαισίας για την πενταετή φυλάκιση του ηγέτου της αντιπολιτεύσεως το Φεβρουάριο φέτος. Ο κύριος Ανουάρ Ιμπραχήμ αρχικά είχε αθωθεί πριν να αντιστραφεί απόφαση, να ανατραπεί απόφαση και ε, εστερήθη των πολιτικών του δικαιωμάτων και έχασε και την έδρα του, την έδρα του βουλευτού. Στις 8 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ε, εταιρική σχέσεως με την Μαλαισία. Επανειλημμένα το Κοινοβούλιο ζήτησε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2011. Αυτή η νέα συμφωνία συμπεριλαμβάνει ειδικέ διατάξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου που θα επιτρέπουν περισσότερη συζήτηση αυτά τα θέματα κυρίως μέσω της δημιουργίας του διαλόγου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις διαπραγματεύσεις η Μαλαισία απεδέχθη να αναγνωρίσει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας. Θα συνεχίσουμε τις επαφές με την κυβέρνηση Μαλαισίας για να αυξηθεί η συνεργασία μας όσον αφορά την προώθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων και των ΛΟΑΔ διμερός καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο με την ΑΖΕΑΝ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Στυλιανίδη. Σας ευχαριστούμε για αυτό το μαραθώνιο της παρουσίας σας που ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Λοιπόν, έλαβα 7 προτάσεις ψηφίσματος τώρα στο ολοκλήρωση συζητήσεως, πέρα συζήτησης. Διακόπτεται η συνεδρία μέχρι τις 12.